Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να δούμε αν έχει να ξεκινάμε δυόμιση. Γιατί οι συνάδελφοι φαίνεται ότι δεν έχουν προσαρμοστεί στα νέα ωράρια. Λοιπόν, να περάσουμε στο σημείο 19 της ημερήσια διάταξης. Έχουμε κοινή συνεδρίαση με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ισομερή Συνέλευση ε, και την αντιπροσωπή μας στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Έχω, δει, έχω εδώ τον ε, Μίχελ Γκάλερ που είναι σύμπροεδρος της αντιπροσωπής μας για το Παναφρικανικό, στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και τον Χουάν Φερνάντο Λόπεθ Αγιλάρ που είναι αντιπρόεδρος της Ισομερούς Συνέλευσης ΑΚΕ ΕΟΚ και θα συμπροεδρεύσουμε. Είναι σημαντικό θέμα. Ο προσκεκλισμένος μας σήμερα το απόγευμα είναι ο πρέσβης Αουατ Σακίμι Αμάντα μόνιμος εκπρόσωπος της ε, Αφρικανικής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος μας είναι να εστιάσουμε στην συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση της, ε, της, της Αφρικανικής Ένωσης. Όπως θυμάστε, ο Πολ Καγκάμε το 2016 επιφορτίστηκε να ετοιμάσει μια έκθεση για την μεταρρύθμιση της Αφρικανικής Ένωσης η οποία κρίθηκε τον ε, Ιανουάριο του 2017 και είναι σε φάση εφαρμογής. Ένα τμήμα αυτής της μεταρρύθμισης είναι η χρηματοδότηση της Αφρικανικής Ένωσης και με βάση τις προτάσεις που εγκλήθηκαν πέρυσι τα μέλη της Ένωσης συμφώνησαν σε ένα σύστημα 2,2% ποσοστού των επιλεξίμων ε, εισαγωγών για να χρηματοδοτηθεί η Αφρικανική Ένωση όπως ακριβώς ε, χρηματοδοτείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω δασμών και τελών. Τον ε, περασμένο Νοέμβρη Πολύ πήγαμε στο Αμπιτζάν στην συνάντηση κορυφής της Αφρικής. Είναι σημαντικό για την ε, Επιτροπή μας προτεραιότητα και χαίρομαι πολύ που είστε εδώ σήμερα κύριε Πρέσβη για να ακούσουμε τη γνώμη σας. Αλλά προηγουμένως να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Λόπεθ Αγγιλάρ που είναι αντιπρόεδρος της ε, Σομερού Συνέλευσης ΑΚΕΟΚ. Ευχαριστώ Λίντα. Καλησπέρα σας. Θα κάνουμε εδώ μία ανταλλαγή απόψεων με τον πρέσβη Αμπάρ Σαχκίλ Αχμέντ για τις σχέσεις μας με την Αφρικανική Ένωση και τη μεταρρύθμισή της. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο φυσικός ε, συνομιλητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και εκπροσωπείται εδώ αυτή η αντιπροσωπεία από τον πρόεδρό μας, τον Μίχαλ Γκάλερ. Ο Λουί Μισελ, ο άλλος συμπρόεδρος, είχε ζητήσει αυτοί οι κοινέ συνεδριάσεις να γίνονται σε μια προοπτική της μετακοτονού εποχής. Η διαπραγματευτική εντολή της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής που ανακοινώθηκε σήμερα φαίνεται ότι καθορίζει την κοινή βάση της σχέσης μας και κυρίως τονίζει τις τρεις περιφερειακές ε, διαστάσεις, συνιστώσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ακόμη πιο στενή σχέση με την Αφρικανική Ένωση και τις ε, περιφερειακές οικονομικές κοινότητες. Γι' αυτό είναι πολύ θετικό το ότι ήδη έχουν προσκαλέσει τους εκπροσώπους της Αφρικανικής Ένωσης στις ε, συνεδριάσεις της Ομερού και ΑΚΕΟΚ και της Ολομέλειας μας. Θεωρούμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ θετικές εξελίξεις ε, στο εσωτερικό της Αφρικανικής Ένωσης. Δημιουργήθηκαν ε, πολλοί θεσμοί και φορείς στα πλαίσια της Αφρικανικής Ένωσης για την ασφάλεια, την καλή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη. Αυτές όμως ε, οι δομές πολλές φορές δεν έχουν επαρκείς πόρους για να ανταποκριθούν ε, στις περιστάσεις. Η έκθεση του κυρίου Καγάμε για την ε, μεταρρύθμιση της Αφρικανικής Ένωσης και του Ντόναλτ Καβελούκα για τη χρηματοδότηση της Αφρικανικής Ένωσης από τα κράτη-μέλη έχουν στόχο να προτείνουν έναν εξορθολογισμό των στόχων και κυρίως να αυξήσουν την οικονομική αυτάρκεια. Ελπίζουμε η παρουσίασή σας, κύριε Πρέσβη, θα μας ε, ενημερώσει για την πορεία εφαρμογής αυτών των δύο εκθέσεων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Φερνάντο, για την εισαγωγή σου. Να δώσω τώρα το λόγο στον Μίχαλ Γκάλα, που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας στο Παναφρικανικό, Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Σε τρεις εβδομάδες θα πάτε, δεν είναι. Ναι, ευχαριστώ, Λίντα. Και ευχαριστώ συνάδελφοι για αυτή την κοινή ανταλλαγή απόψεων και εγώ να καλωσορίσω θερμά τον πρέσβη που συμμετείχε στις 5 Μαρτίου στη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας μας. Όπως είπε ο συμπρόεδρος της ε, συνέλευσης, ΑΚΕΟ, Λουί Μισελ είπε, διαπραγματεύσεις για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ των χωρών Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όπου συμμετέχουν 48 αφρικανικές χώρες. Και βεβαίως το Μάιο θα επισκεφθούμε το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και εκεί θα συζητήσουμε τις επιπτώσεις της μετακοτονού εποχής. Στις συνεδριάσεις της κοινή ε, ισότιμης συνέλευσης πάντα τονίσαμε την κοινοβουλευτική διάσταση των μελλοντικών αυτών σχέσεων. Γιατί αυξάνεται η σημασία της περιοχής αυτής και γι' αυτό καλό τώρα να μεταρρυθμιστούν αυτοί οι θεσμοί και ρωτάω εάν προβλέπουν και ενίσχυση του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και πώς θα εφαρμοστεί συγκεκριμένα και πότε. Βεβαίως, επίκειται η ενίσχυση του καταστατικού του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου που θα του επιτρέψει να περάσει κάποια πρότυπα νομοθετήματα ως προτάσεις για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το στάδιο, γιατί πρέπει να υπογραφεί, να επικυρωθεί από όλες τις χώρες και άρα η έναρξη ισχύω απέχει ακόμη πολύ. Οπότε γι' αυτό τίθεται και το ερώτημα θα υπάρξουν άλλες γενικότερες μεταρρυθμίσεις ή αυτέ θα είναι και θα είναι ιδιαίτερα μακρόπνοη η διαδικασία χωρίς να μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα αρχίσει να ισχύει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και πρόεδρος. Πολλές ερωτήσεις πριν καν πάρετε το λόγο, αλλά σα δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές που είναι παρόντες και για να σας δείξω ακόμη μια φορά τη διάθεση της Αφρικανικής Ένωσης ε, για ανταλλαγές απόψεων και επίσης ε, και για μας είναι σημαντικές και αποδεικνύει και το ενδιαφέρον που ε, αποδίδουμε και εμείς σε αυτή τη συνεργασία. Θα ήθελα καταρχάς σε σχέση με το θέμα που είναι στην ημερήσια διάταξη της μεταρρυθμίσης, πρόκειται για τις μεταρρυθμίσεις της Αφρικανικής Ένωσης. Όπως το γνωρίζετε, είναι σημαντικό δεδομένο για τους Αφρικανούς ηγέτες. Μετά από την Αφρικανική Ενότητα, η Αφρικανική Ένωση ε, ήταν η εξέλιξη αυτής, αλλά θα πρέπει να οδηγηθούμε και σε μια περαιτέρω μεταρρύθμιση που θα καταστήσει την Αφρικανική Ένωση και του θεσμού της αποτελεσματικούς και υποθετικού. Να είμαστε πιο λειτουργικοί δηλαδή. Έχουμε μπει σε μια σταδιακή μεταρρύθμιση και όπω γνωρίζετε όλη η διαδικασία ξεκίνησε τον Ιούλιο 2016. Έλεγα μάλιστα ότι πρόκειται για μια ιστορική μέρα για την Αφρικανική Ένωση, διότι τότε ξεκίνησε όλη η μεταρρύθμιση στο Κιγκαλί ε, με την 27η διάσκεψη κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης, όπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν να αναθέσουν τη μεταρρύθμιση στον πρόεδρο Καγκάμε. αυτή απο... Ε, αποστολή λοιπόν έχει ως στόχο να καταστήσει πιο αποδοτική και παραγωγική τη λειτουργία των διαφόρων οργάνων της Ένωσης. Ήταν επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της Ένωσής μας και γι' αυτό το λόγο μια από τις προτεραιότητες που διαγράφονται από αυτή την έκθεση, κάποιες μάλλον προτεραιότητες είναι η εξή. Πρέπει να τονιστούν οι, προτεραιο, οι προτεραιότητες κλειδιά, πράγμα που θα επιτρέψει επίσης σε επίπεδο της ε, μεταρρύθμισης ε, Πρόκειται για τις πολιτικές υποθέσεις, όπως γνωρίζετε, εκεί έχουμε μια μεγάλη αρχιτεκτονική για τη διακυβέρνηση και τις εκλογές που και εσείς υποστηρίζετε μέσω της καθοριστικής στήριξης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, μας απασχολεί και απασχόληση. Το 85% των ενόπλων σειράξεων ε, ε, σοβούν στην Αφρική. Πράγμα το οποίο μας κάνει να προβληματιστούμε για να ενισχύσουμε τη συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στο Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης καθώς επίσης και το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ευρώπης και χωρίς να ξεχνάμε και την πολυμερή συνεργασία ε, που υπάρχει με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε επίσης την οικονομική ολοκλήρωση. Η οικονομική ολοκλήρωση ε, μια υπήρου που αποτελείται από 55 κράτη θα πρέπει να δούμε πώς ας πούμε, θα μπορέσουμε να έχουμε την ε, κινητικότητα στην Αφρική, τη δυνατότητα εγκατάστασης, αλλά και να δημιουργήσουμε και μια ε, πανυπηρωτική ε, ζώνη ελευθέρων συναλλαγών που θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, που είναι ένας από τους πρώτους εταίρους της των Αφρικανικών χωρών. Αυτό τονίστηκε στην τελευταία διάσκεψη κορυφής στο Αμπιτζάν να έχουμε δηλαδή ενισχυμένη συνεργασία και έτσι να ενισχύσουμε και τις εμπορικές σχέσεις αλλά και να αναχαιτήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης. Μια άλλη πτυχή που καλύπτεται είναι πώς και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να ακουστεί η φωνή της Αφρικής σε διεθνές επίπεδο. Όπως γνωρίζετε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ που είναι εκείνο που αποφασίζει με τα πέντε μόνιμα μέλη του, όμως ο κόσμος έχει ε, εξελιχθεί σε επίπεδο συγκρίσεων, όπως σας έλεγα, 80% των ε, ενόπλων σειράξεων σοβούν στην Αφρική, οπότε είναι αδιανόητο να λειτουργεί μόνο με πέντε μέλη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να μπορεί να αποφασίζει ε, για την ασφάλεια μόνο το αυτό για, για την Ευρώπη, για, ε, για την Αμερική, την Λατινική Αμερική. Ε, πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με την Ευρώπη μέσα στο πλαίσιο της εντολής των μη μονίμων μελών, των, των Ευρωπαίων μελών, που πάντοτε είχαν τη στήριξη την καθοριστική της Αφρικής. Πάντοτε συνεργαζόμαστε σε αυτά τα θέματα. Να θυμίσω όπως ξέρετε η Αφρικανική Ένωση αποτελείται από διάφορες επιτροπές. Έχουμε 8 επιτροπές. Έχουμε και 11 όργανα με 20 επιτροπές και υποεπιτροπές και επιτροπές υψηλού επίπεδου διεπουργικές αλλά και ε, επιτροπές ε, όπως αυτή προσανατολισμού που αποτελείται από ηγέτες και αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων είναι και ένα όργανο που έχουμε το ΝΕΠΑΝΤ. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης θα γίνει ένα εκτελεστικό ε, φορέας, αντί να είναι ένας θεσμός ξεχωριστός. Θα ε, συνδεθεί με την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης και θα διαχειρίζεται τα project προτεραιότητας που περιλαμβάνονται ε, στο θεματολόγιο μας. Οδηγηθήκαμε λοιπόν στο να ξεκινήσουμε αυτή τη μεταρρύθμιση λαμβάνοντας υπόψη το, τα όσα υπάρχουν στην ατζέντα μας, γιατί στην Αφρική δεν έχουμε ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα. Ας πούμε σε 50 χρόνια αυτοί που θα είναι τότε εκεί θα το δουν. Έχουμε και ένα μηχανισμό αξιολόγησης από τους εταίρους μας, από τους ομολόγους μας, ώστε ας πούμε να τονιστεί η διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα από το χαμηλότερο μέχρι το ψηλότερο ώστε να δούμε πώς σε επίπεδο χωρών τα διάφορα όργανα και οι διοικήσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργούν. Στόχος είναι να υπάρχει λογοδοσία Σε σχέση τώρα με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, που ο ρόλος του μέχρι στιγμής είναι συμβουλευτικός, και εκεί υπάρχει εξέλιξη προς ένα κοινοβούλιο που σύντομα θα έχει και νομοθετικές ε, αρμοδιότητες γιατί και πολύ σημαντικό γιατί όπως γνωρίζετε ολοκλήρωση είναι πολύ μακρά πορεία ε, αν σκεφτείτε την ευρωπαϊκή ιστορία ξεκίνησε πολύ νωρίτερα και συνεχίζεται η ενίσχυση του Κοινοβουλίου. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να έχουμε ένα Κοινοβούλιο πιο αντιπροσωπευτικό, με πιο εκτεταμένες άξιες αρμοδιότητε, αρμοδιότητες, πράγμα το οποίο αποφασίστηκε στο Μάλαμπο ε, με σχετικά πρωτόκολλα κτλ. Θέλουμε επίση να προσεγγίσουμε του πολίτε στην Αφρικανική Ένωση. Πρόθεση ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι μια αρχή που περιλαμβάνεται στο καταστατικό της Αφρικανικής Ένωσης. Έχουμε θεσπίσει στόχους ε, για την ισότητα ανδρών γυναικών. Δεν υπάρχουν θέσεις απασχόλησης που να ε, μην μπορούν να προσληφθούν γυναίκες. Η Αφρικανική Ένωση είναι πραγματικός και υπερασπιστής της ισότητας. Γι' αυτό και στην ε, Κομισιόν έχουμε δημιουργήσει ένα όργανο που ασχολείται ήδη με την ισότητα και έχουμε ενισχύσει και τις δυνατότητες των γυναικών, γιατί είδαμε την αποτελεσματικότητα των γυναικών όσον αφορά την διαμεσολάβηση σε χώρες που βρίσκονται σε σύραξη. Να θυμίσω λοιπόν, ήθελα να θυμίσω τους στόχους, μέχρι το 2025 θέλουμε να αυξηθεί και η ποσόστοση των νέων, γιατί οι νέοι είναι στη βάση όλων, γιατί η Αφρική είναι μια πολύ νεαρή ήπειρος, έχουμε πάρα πολλούς νέους και όσο πάει θα αυξάνονται. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, θα πρέπει να επιταχυνθεί. Οι γυναίκες βρίσκονται στη ε, μέτωπο για όλη αυτή τη διαδικασία και θέλουμε να ενισχύσουμε και τις δραστηριότητες του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου ώστε να υπάρχει επιστοποίηση της κοινωνίας των πολιτών ώστε και αυτή να είναι φορέας της ανάπτυξης και να συμμετέχει στη δραστήρια ζωή σε επίπεδο των οργάνων της Αφρικανικής Ένωσης. Ένα άλλο στοιχείο είναι η χρηματοδότηση της Αφρικανικής Ένωσης με βιώσιμο τρόπο. Όπως αναλάβαμε, καθώς αναλάβαμε την δέσμευση να ε, ακολουθήσουμε το Agenda 2063 με το πρώτο δεκαετές πρόγραμμα, θα πρέπει η Αφρική να περιμένει μέχρι ότου οι εταίροι να χρηματοδοτούν την ανάπτυξή της. Γι' αυτό και δεσμευτήκαμε να ε, χρηματοδοτήσουμε 100% τις λειτουργικές δαπάνες της Αφρικανικής Ένωσης, δηλαδή συντήρηση κτίριων, ε, αμοιβές ε, του προσωπικού, αλλά και τις δραστηριότητες ε, που έχουμε στο πρόγραμμά μας και 25% να καλύψουμε τα κονδύλια για την ειρήνη και την ασφάλεια. Διότι διαπιστώσαμε με το πρόγραμμα της εφαρμογής της ε, αφρικανικής ε, δύναμης για την άμεση αντίδραση στις κρίσεις θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις παρέμβασης. Όταν ας πούμε ξεσπά μια ε, σύγκρουση κάπου θα πρέπει να μπορούμε να αντιδράσουμε άμεσα πριν γίνει καταστροφική κατάσταση. Θέλουμε λοιπόν μέσω αυτού του Ταμείου για την Ασφάλεια να έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να μπορούν γρήγορα να παρέμβουν ε, θετικέ δυνάμεις. Όπως έγινε, θα το είδατε με την ε, ε, δύναμη που συστάθηκε από τους G5 Σαχέλ. Εκεί δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να υπάρχουν αυτά τα κονδύλια έτοιμα. Αλλά να στηρίξουμε και με τα κονδύλια του ΟΗΕ σε περιπτώσεις ε, ε, ασφάλειας για το υπόλοιπο 75%. Να θυμίσω επίσης τον φόρο 0,2% Έχουμε τον ε, Κάρλος Κάρλος που ήταν ο Γενικός Γραμματέας ε, της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Αφρική 0,2% για όλες τις εισαγωγές. Επιβάλλεται φόρος για όλες τις ε, εισαγωγές που είναι φορολογητές. Βέβαια, λαμβάνοντα υπόψη όλες τις συμφωνίες ε, οικονομικής εταιρική σχέσης που έχουμε με τους συνεργάτες μας, με τους εταίρους μας, να μπορούμε λοιπόν να συλλέγουμε αυτό το φόρο, πράγμα που θα επέτρεπε να λειτουργήσουμε. Σας διαβεβαιώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, ότι τα πράγματα προχωρούν. Γιατί για πρώτη φορά έχουμε αρκετά σημαντικό αριθμό χωρών που συμμετέχουν. Το Ταμείο για την Ειρήνη και την Ασφάλεια επίσης έχει πρικοδοτηθεί και συνεχίζουμε παρότι υπάρχουν δυσκολίες Γι' αυτόν τον λόγο δημιουργήσαμε μια Επιτροπή Υπουργών Οικονομικών και Υπουργών Εξωτερικών, 15 υπουργοί, έχουμε πάρει τις διάφορες ε, περιφέρειες, ώστε να ε, τελειοποιήσουμε και να ολοκληρώσουμε την εξέταση αυτών των θεμάτων. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συμφωνίες που υπάρχουν και να μην εκμεδενήσουμε τις προσπάθειες και τις δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει απέναντι στου εταίρου μα εδώ λοιπόν τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Επίσης, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης ήθελα να σας δώσω συγκεκριμένα ε, ε, ενέργειες, Το έναρξη της ζώνης ελευθέρων συναλλαγών που ε, άρχισε να ισχύει, μάλλον τη δέσμευση που αναλάβαμε στις 20 Μαρτίου στο Κιγκαλί. Θα έχουμε συνεργασία ελευθέρων συναλλαγών με ένα πλάνο και θα σας το υπεβάλλουμε, θα σας το παρουσιάσουμε, καθώς και ένα πρόγραμμα εκβιομηχανισμού. Θέλουμε να έχουμε μια εκβιομηχανισμένη Αφρική άνευ συνόρων και μια Αφρική που θα είναι ανοιχτή προς την Ευρώπη, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ε, ε, εταίρους μας. Υπάρχει δυνατότητα σε όλους τους ευρωπαίους οικονομικούς φορείς να έρθουν να επενδύσουν στην Αφρική σε όποιον τομέα θέλουν. Όμως, επίσης, να έχουμε και εμπόριο ένδοαφρικανικό ανάμεσα στις χώρες. Ε, έχει επίσης, υπάρχει το δικαίωμα αποζημίωσης ε, που θα βοηθήσει στις ε, εμπορικές αναλλαγές, αλλά και το δικαίωμα του διαβατηρίου. Πάλι στο Κιγκαλή αυτό θεσπίστηκε. Μαζί με το Ευρωπαϊκό ε, ε, διαβατήριο μπορεί κανείς να φύγει από τη Λιβύη και να βρεθεί στη Νότια Αφρική, από τη Ζιμπάμπο να πάει στο Μαρόκο και ούτω καθεξής. Θέλουμε δηλαδή μέσω ε, της δικής του δικού σας σώματος να μπορέσουμε και εμείς να θεσπίσουμε αυτό, αυτό το, την Αφρανική Ένωση Βεβαίω έχουμε υπόψη ότι έχετε και εσείς τις υποχρεώσεις σας εννοείται, το γνωρίζουμε. Ε, θέλουμε μέσα στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου να μπορέσουμε να οργανωθούμε για να ρυθμίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Μια άλλη πτυχή που έχουμε επίσης ε, θίξει, κυρία Πρόεδρε, ε, έχουμε τα, την μεταρρύθμιση αλλά και τα προγράμματα 2020, δηλαδή τις διαπραγματεύσεις για το Κοτονού, τη Συμφωνία Κοτονού μετά το 2020. Μετά από την μελέτη που έγινε από την Ευρώπη, νομίζω πως έχει δημοσιευθεί το Δεκέμβριο του 2017 και στο επίπεδο της Αφρικής έχουμε σκεφτεί, έχουμε προβληματιστεί λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς και τις κατευθύνσεις που προέκυψαν από τη διάσκεψη κορυφής του Αμπιτζάν. Θέλουμε να έχουμε σχέσεις μετα... ίσο προς ίσο. Όχι σχέσεις μεταξύ εταίρου και δωρητών. Εταίρων και δωρητών. Αυτό νομίζω ε, το ακούσατε και στην ε, Ολομέλεια του Στρασβούργου από τον πρόεδρο που βρέθηκε εκεί. η απόφαση νομίζω που ελήφθη σχετικά στο Κιγκαλί έχει δημοσιευθεί, πράγμα που θα επιτρέψει στην Αφρική να λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα. Υπάρχουν δεσμεύσεις που, για την Βόρεια Αφρική που ε, ε, θα διατηρηθούν, αλλά και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει μέσα στο πλαίσιο των ενδεικτικών εθνικών προγραμμάτων, αλλά και στο πλαίσιο των περιφερειακών ε, προγραμμάτων. Θέλουμε λοιπόν να μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα σε Ένωση και Ένωση και Ήπειρο και Ήπειρο, λαμβάνοντας υπόψη όμως και όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν από κοινού, τις κλιματικές αλλαγές ας πούμε, με την Ευρώπη είχαμε ανέκαθεν ε, κοινέ θέσεις, πράγμα που έχει επιτρέψει στην Αφρική και στην ε, Ευρώπη να στηρίξουμε την Ατζέντα 2030, αλλά και την κοινή, ε, οι κοινέ αυτές θέσεις δίνουν νέα όθηση για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε συνεργασίες, συνεργασίες με την Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Η Αφρική έχει εταιρική σχέση με την Ευρώπη, με τις και με την Τουρκία αλλά και με την Ινδία και τον αραβικό κόσμο. μέσω αυτών των κυκλικών σχέσεων που έχουμε και των ιστορικών σχέσεων που έχουμε με την Καραϊβική και τον Ειρηνικό, η απόφαση του ε, Συμβουλίου μας ε, δίνει τη ε, δικαιοδοσία στους υπουργούς να διαπραγματευτούν συμφωνία συνεργασίας με την Καραϊβική και τον Ειρηνικό θα τελειοποιήσουμε την κοινή μας θέση, πράγμα το οποίο θα δώσει τη θέση του σε μια διαπραγματευτική ομάδα όπως και στην Ευρώπη και την κατάλληλη στιγμή ελπίζω πως θα μπορέσουμε να συνοηθούμε ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε ε, καρποφόρα αυτή τη σχέση. Η κοινή αφρικανική θέση που έχει ε, θεσπιστεί θα επιτρέψει να έχουμε συνεδριάσει σημαντικές ανάμεσα στους Υπουργούς Εξωτερικών από Ήπειρο σε Ήπειρο πράγμα που θα επιτρέψει ανταλλαγές ε, ε, πολιτικού και διπλωματικού επίπεδου, χωρίς να ξεχνάμε και τις επαφές ανάμεσα στην Κομισιόν, κάθε φορά Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης, αλλά να δούμε και πώς τα κοινοβούλια θα μπορέσουν να βελτιώσουν ε, τις επαφές τους και τη συνεργασία τους, δεδομένου ότι και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο προσεχώς θα είναι αντιπροσωπευτικό. Έχουμε προβλέψει και διπουργικές ε, συσκέψεις στο πλαίσιο του εμπορίου, της παιδείας, της υγείας, έτσι ώστε οι Αφρικανοί υπουργοί να μπορέσουν να συζητήσουν με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους για αυτά τα θέματα, όπως και για τη μετανάστευση. Να δούμε πώς εξελίσσεται η διαδικασία της Βαλέτας, της Χαρτούμ, του Ραμπάτ, ε, πώς με όλα αυτά τα κεκτημένα σε επίπεδο της Βόρειας Αφρικής θα, μπορέσουμε, θα μπορέσουν να ωφεληθούν και οι υπόλοιπε αφρικανικές χώρες. Ξέρουμε πώς, δεσμευτικά είναι, πώς είναι δεσμευτικές αυτές οι συμφωνίες. Το, το παράδειγμα τους όμως θα μπορούσε να ωφελήσει και τα άλλα κράτη της Αφρικανικής Ένωσης αλλά και Τις συνεργα... συνεργασία συνεργασίας με τη ΣΑΔΕΚ είναι πράγματα που υπάρχουν και που θα ενισχυθούν και θα ε, επεκταθούν και στις άλλες χώρες, έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε ιστορικές συμφωνίες μεταξύ μας. Δεν θα πρέπει να σκεφτείτε ότι η Αφρική ε, εγκαταλείπει την Καραϊβική και τον ε, Ειρηνικό. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε όμως να υπάρχει συνοχή ανάμεσα ε, στα δικά μας project ολοκλήρωσης. Η Ευρώπη θα μπορέσει να συνεργαστεί και με τις περιφερειακές οικονομικές ενώσεις που υπάρχουν, μάλλον επιτροπές που υπάρχουν. Αυτά είχα να σας πω και αυτά προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση αλλά και από το φιλόδοξο πρόγραμμα που ε, σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε. Υπάρχει και ένα project το οποίο είναι επίσης εξίσου σημαντικό είναι η ενιαία αγορά των αεροπλοείας των αεροπορικών μεταφορών. Η Αφρική έχει ανοίξει τον εναέριο χώρο τη σε όλες τις εταιρείε Θα έχουμε θεματικές συνεδριάσεις και τεχνικές επίση συνεδριάσεις ώστε να ανοίξει ε, πραγματικά ο εναέριο χώρο μας, πράγμα που θα επιτρέψει σε όλες τις εταιρείε να έχουν πρόσβαση στον αφρικανικό ουρανό και άρα να έχουμε ακόμα περισσότερες συναλλαγές. Κυρίως βασιζόμαστε πολύ στην Ευρώπη ώστε αυτό το σημαντικό project να ε, φτάσει σε αίσιο πέρας. Αυτά, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι Ευρωβουλευτές, αυτές είναι οι πληροφορίες που επιθυμούσα να μοιραστώ μαζί σας ώστε να μπορέσουμε μαζί να συνομιλήσουμε, να, να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Πράγματι είναι φορτωμένη η ατζέντα σας καθώς και φιλόδοξο το πρόγραμμα για την Αφρικανική Ένωση. Και είμαι βεβαία ότι αυτό, αυτά θα ενδιαφέρουν πολύ τους συναδέλφους. Πριν τους δώσω όμως τον λόγο στους συναδέλφους, θέλω να τονίσω ότι έχουμε ορισμένου προσκεκλημένους εδώ μεταξύ μας από την Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, τον κύριο Μαλεόμπο, επικεφαλής του, ιδιωτικού, του προσωπικού γραφείου του αρχηγού του κράτους, τον κύριο Ορομφέ, που είναι επίσης αρμόδιος για τις νέες τεχνολογίες για τον Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Επίσης, να πω το εξής. Χθες στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή συζητήσαμε τις σχέσεις με την Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, διότι όσο θα γνωρίζετε, κάποιοι από εμά επισκεφθήκαμε την χώρα σας τον Μάρτιο. Και είχαμε την τιμή να μας δεχτεί ο ίδιος ο πρόεδρος σας, καθώς και ο Πρωθυπουργό, ε, με τους οποίους προέβημεν σε πολύ χρήσιμες ανταλλαγές απόψεων. Και επανήλθαμε εδώ με το μήνυμα της ανάγκης ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Κάποια πρόοδο έχει γίνει στι σχέσει αυτέ, αλλά μένει ακόμα πολύ δουλειά να γίνει και τη δουλειά αυτή πρέπει να την αναλάβουμε από κοινού. Θέλουμε να ενισχύσουμε τι σχέσει με το κοινοβούλιο σα, με του βουλευτέ σα, Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα ικανοποιημένη που είστε σήμερα παρόντες εδώ και μπορείτε να συμμετάσχετε στην συζήτηση για την Αφρικανική Ένωση. Στις 3.30 θα αναγκαστώ να αποχωρήσω από την αίθουσα, αλλά ο συνάδελφός μου και αντιπρόεδρος κ. Ντέβα θα με αντικαταστήσει και είμαι βέβαιος ότι εάν επιθυμείτε να λάβετε το λόγο θα σας τον δώσει. Έχει καλώς. Τώρα, ποιο θα ήθελε να λάβει το λόγο, κυρία Ντονανό. σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξοχότατε κύριε ε, μόνιμη εκπρόσωπε, μόνιμη αντιπρόσωπε. Ο διάλογος θα είναι αμοιβαία αποφελής, ελπίζω, για τις Ευρωπαϊκέ και για τις αφρικανικές γόρες. Για τους τρεις πυλώνες που είναι η ανάπτυξη, η πολιτική, η η πολιτική, η οικονομία και το εμπόριο, οι προσπάθειες θα βασιστούν στους πυλώνες που είναι προτεραιότητα για την Αφρική, μετανάστευση, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, δικαιώματα ανθρώπου και η διαχείριση των φυσικών πόρων. Ως γνωρίζετε, η μεταναστευτική κρίση μπορεί να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να είναι απαιτητικότερη σε ό,τι αφορά επανεισδοχή και επιστροφή απέναντι στους εταίρους της ε, του ε, Νότου. Ε, δεν είναι δυνατόν να διδαχθεί κανείς στην μετανάστευση, ωστόσο, εάν δεν αντιμετωπίσει τις ρίζες της. Η ερώτησή μου λοιπόν έχει ως εξής. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος κατά την άποψή σας για να στηρίξουν την απασχόληση οι χώρες μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις χώρες εταίρους τους. Και εάν οι στόχοι αυτοί αποτελούν μια καλή βάση, πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε τον πολλαπλασιασμό αυτών των πυλώνων και των φιλοδοξιών, που τελικώς ενδέχεται να οδηγήσουν σε ματαιώση των προσπαθειών. Σας ευχαριστώ για την απάντηση που θα δώσετε. Ο Μιχαήλ Γκάλερ, ευχαριστώ έχω πράγματι εντυπωσιαστεί από το φιλόδοξο πνεύμα που απηχούν τα κείμενα και αποφάσεις που λαμβάνει η Αφρικανική Ένωση. Αναφέρεστε σε ένα διαβατήριο της Αφρικανικής Ένωσης. Αρκεί αυτό να μην σημαίνει ένα ακόμη διπλωματικό διαβατήριο για κάποιους Αφρικανούς διπλωμάτες, αλλά θα πρόκειται για ε, διαβατήριο το οποίο θα επιτρέπει σε Αφρικανούς πολίτες να μεταβαίνουν από τη μια χώρα στην άλλη. κατάλαβα καλά ότι κάποια στιγμή το ταξίδι εντός Αφρικής ε, θα είναι απαλλαγμένο της υποχρέωσης προξενικών θεωρήσεων και προβλέπετε κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα ή θα το καθορίσετε βήμα προς βήμα μεταξύ των χωρών οι οποίες ήδη έχουν τις ρυθμίσεις αυτές μεταξύ των και θα διευρυνθεί σιγά σιγά ή εν πάση περιπτώσει πώς σκέπτεστε να προχωρήσετε. Για την καθιέρωση Παναφρικανικού χώρου ελευθέρων συναλλαγών. Όσο γνωρίζουμε όλοι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ενοποίησης σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές υπάρχουν ήδη τελωνιακές ενώσεις. Για να φτιάξετε λοιπόν τώρα ένα παναφρικανικό χώρο ελευθέρων συναλλαγών, αυτός θα βασιστεί σε υφιστάμενα project που υπάρχουν ήδη, δηλαδή ή θα αρχίσει από το μηδέν και θα δείτε πού μπορείτε να συμφωνήσετε σε, κάποια, σε κάποιους κοινούς δασμούς ή πρότυπα που μπορούν να υιοθετηθούν ή πώς αλλιώς να φανταστούμε την εφαρμογή στην πράξη αυτού του μεγαλεπίβολου σχεδίου. Ευχαριστώ. Έκρεψε την ερώτησή μου για τα διαβατήρια. Νόρμπερτ Νόρισερ. ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ για την ανάπτυξη του φιλόδοξου αυτού προγράμματος που εξηγήσατε, ερώτηση σχετικά με τις σχέσεις με ταξί των χωρών ΑΚΕ, Αφρικής Καραβικής Ειρηνικού. Βρισκόμαστε τώρα στα προεόρτια της ε, συμφωνίας μετά την Κοτονού έχουμε δύο διαφορετικούς μορφότυπους τώρα για την Αφρική. Αφενός τη σχέση μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη μεριά ε, το αν θα περιληφθούν οι χώρες ΑΚΕ. Δεν είναι και τόσο διαρθρωμένα αυτά όσο κάποια άλλα σχέδια γιατί οι, Αφρικα... οι βόρειο αφρικανικές χώρες δεν εντάσσονται στην ε, κοινότητα των χωρών ΑΚΕ θα ενταχθούν ή πώς θα το διαχειριστείτε αυτό στο μέλλον, γιατί υπάρχουν δύο επικαλυπτόμενες δομές. Και θα ήταν καλό να διαρθρωθεί καλύτερα η σχέση μεταξύ του συνόλου της Αφρικανικής Υπήρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη, θα θέλατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου σχετικά με την ερώτηση για τους πυλώνες που διατηρούνται στην κοινή αφρικανική θέση. Σας διαβεβαιώ ότι οι πυλώνες αυτοί περιλαμβάνονται έχουν επιβεβαιωθεί και από, το πρόσφατο, από την πρόσφατη διάσκεψη κορυφής Αφρικανικής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί περιλαμβάνεται και η απασχόληση. Για το θέμα της μετανάστευσης έχω μια προσωπική άποψη αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν θα μπορέσει να ρυθμιστεί το θέμα της μετανάστευσης εάν, εάν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στις ε, βαθιές του ρίζες διότι οι Αφρικανοί ρίχνονται σε μια περιπέτεια για να έρθουν να βρουν το Ελτοράδο τους εδώ στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί. Όχι μόνο μέσα της απασχόλησης. δεν θα μπορέσει να δοθεί απασχόληση στον κόσμο εάν δεν εκβιομηχανιστεί η Αφρική. Χρειάζεται λοιπόν μια βιομηχανική πολιτική, να δημιουργηθούν βιομηχανίες και να προσληφθεί το ανθρώπινο αυτό εργατικό δυναμικό, το οποίο είναι ακόμη νεαρό σε ηλικία και έχει ε, φιλοδοξίες, σχέδια και ελπίδες. Δηλαδή χρειάζεται να γίνει αυτό για να δημιουργηθεί απασχόληση. Για την μετανάστευση, επανεισδοχές, επιστροφές, προξενικές θεωρήσεις κλπ. Όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει με την Ευρώπη, το θυμούμε καλά και συνεχίζουμε να τα συζητούμε. Αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό κάπως συνεκτικό. Έχουμε ένα πλήθος υφιστάμενων μηχανισμών, της βαλέτας, του χαρτούμ, του ραμπάτ. Μηχανισμοί οι οποίοι λειτουργούν, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να καθίσουμε να αξιολογήσουμε πώς λειτουργούν τα προβλήματα της μετανάστευσης. Δεν είναι μονάχα αφρικανικά προβλήματα. Και στην Ευρώπη έχετε το ίδιο πρόβλημα. Πώς μπορούμε εμείς να επωφεληθούμε στην Αφρική από την εμπειρία σας και να κάνουμε ανταλλαγή εμπειριών για να μπορέσουμε από κοινού να λύσουμε το πρόβλημα. Για να λύσουμε το πρόβλημα τη κινητικότητα των ανθρώπων, δίνοντα προξενικέ θεωρήσει σε αυτού που πηγαίνουν να βρουν δουλειά. Και αυτοί που δεν είναι νόμοι να επαναπατριστούν. Πώ να επαναπατριστούν και να έχουν οι άνθρωποι αυτοί δουλειά στους, στον τόπο του για να μην προσπαθήσουν να επιστρέψουν εδώ. Για το θέμα που τέθηκε για το ερώτημα μάλλον του Παναφρικανικού χώρου ελεύθερων συναλλαγών. Θέλουμε μέσα στην Αφρικανική Ένωση να φτιάξουμε ένα χώρο ελεύθερων συναλλαγών. Αυτό ήταν και το πρώτο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να κάνει κανείς μια ένωση οικονομική ή νομισματική εάν έχει προτιμησιακούς δασμούς. Και υπάρχουν προτιμησιακοί δασμοί στη βάση των οικονομικών συμφωνιών που έχουμε με την Ευρώπη στα πλαίσια, για παράδειγμα, των περιφερειών που λειτουργεί, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς αξιολογούνται οι συνεργασίες αυτές. Να έχουμε ένα νήμα το οποίο θα διέρχεται μέσα από όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Όχι 14-15 προτιμησιακούς δασμούς, αλλά που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να έχει κάποια πλεονεκτήματα, αλλά αυτά κινδυνεύουν να κατακαιρματίσουν τις προσπάθειες. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να ενισχυθούν τα κεκτημένα για να μπορέσει να υλοποιηθεί ο χώρος ελεύθερων συναλλαγών. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της κατάστασης μετά την Συμφωνία Κοτονού, γνωρίζετε κι εσείς όπως και εμείς όλοι είμαστε πεπισμένοι ότι χρειάζεται μια αναθεώρηση των υφισταμένων συμφωνιών. Εάν πάρουμε σήμερα την Αφρική όπως, είναι, όπως έχει σήμερα. Έχουμε μια Αφρική η οποία έχει συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Υπάρχει το ΣΑΝΤΕΚ. Έχουμε τις 48 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Και μετά τη διάσκεψη του Αμπιτζάν είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σχέση μεταξύ των δύο υπήρων. Αυτό επιζητούμε. Η Ευρώπη επιζητά την περιφερειοποίηση. Αυτό και σε εμά. Ωστόσο, καλύτερα να συνεργαστεί ένωση με ένωση, διατηρώντας τα είδη και εκτιμένα. Και την Αφρική του ΣΑΝΤΕΚ, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα ενδεικτικά εθνικά προγράμματα και τα ενδεικτικά περιφερειακά προγράμματα. Πώς θα αντιμετωπιστούν τώρα όλα αυτά, των πολυμερών σχέσεων μέσα στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών. Αυτό όμως θα επιτρέψει να ενισχυθεί και ο διάλογος. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία που να πάρει ένα μέρος της Αφρικής και να το κολλήσει στην Καραϊβική. Αυτό δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της απόφασης που λήφθηκε. Χρειαζόμαστε μια κοινή θέση που να εξετάσει το σύνολο των 50 τόσων χωρών φτιάχνοντας μια αρχιτεκτονική θεσμική δομή που θα επιτρέψει την διαχείριση της υπόθεσης αυτής. Με την Καραβική και με τον Ειρηνικό έχουμε κοινά σημεία τα οποία αντιμετωπίζουμε για παράδειγμα κλιματικής αλλαγής. Έχουμε και σχέσεις φιλικές και αίματος που μας συνδέουν. Θέλουμε όμως ένα, μια ξεχωριστή συμφωνία. Και η Georgetown έδειξε τις ε, τα όρια της. Παρόλο που έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη. Υπάρχει όμως τρόπος να αντιμετωπιστεί μια κατακαιρματισμένη Αφρική στη σχέση της με μια ενωμένη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια ενωμένη Αφρική η οποία να μιλεί με μια φωνή, να έχει κοινέ θέσεις, κάτι που θα επιτρέψει και στον εταίρο μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να επωφελθεί από τα πλεονεκτήματα που ε, προσφέρουμε. Και αυτό να είναι αμοιβαίο. Απάντησα, κύριε Πρόεδρε, στις ερωτήσεις που μου έθεσαν οι αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Ναι, ναι, πολύ καλά. Ο κύριος Γκέρνς θέλει να πει κάτι ακόμη. Σας παρακαλώ να είστε σύντομος. Γιατί πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Παρακαλώ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Εντυπωσιαζόμεθα από τις ε, προόδους που έχουν σημειωθεί και που είναι οσιώδεις σε διάφορες ε, πλευρές στην Αφρική. Αλλά πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν. Πρώτα απ' όλα στον τομέα της ασφάλειας. Όντως η Αφρικανική Ένωση έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Αλλά από πλευράς διακυβέρνησης δεν πάνε τόσο καλά τα πράγματα. Για παράδειγμα, δεν εκπροσωπείται σωστά η Αφρική στα Ηνωμένα Έθνη. Θα έπρεπε να αποδοθεί μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θα πρέπει να δοθεί στην Αφρικανική Ένωση. Και η Αφρικανική Ένωση θα μπορούσε να ορίσει τον εκπρόσωπο της Αφρικής. Και δεύτερον, καθυστέρησα λίγο, δεν ξέρω αν ασχοληθήκατε με τις σχέσεις Αφρικής-Κίνας η Κίνα παίζει μεγάλο ρόλο στην Αφρική. Πώς αξιολογείται το ρόλο της. Τα πρότυπα ανάπτυξη, τα πρότυπα συνεργασία είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ ημών και της Κίνας. Εμείς ως Αφρική ε, θέτουμε προϋποθέσεις. Πολύ έντονες. Οι οποίες περιλαμβάνονται και στις συμφωνίες μας με την Αφρική. Ενώ η Κίνα έχουμε την εντύπωση ο μόνος όρος που έθετε είναι να μην αναγνωρίζουν οι αφρικανικές χώρες την ε, Ταϊβάν. Σήμερα δεν έχουμε ιδέα. Αυτές οι δύο τόσο διαφορετικές ε, αντιλήψεις ε, αλληλοσυμπληρώνονται ή αλληλοαποκλείονται. Σας παρακαλώ πολύ σύντομα κύριε Πρέσβη γιατί να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ω Αφρικανική Ένωση έχουμε πολλές εταιρικέ σχέσει μεταξύ τη οποία και η συνεργασία μας με την Κίνα. Στόχο μα είναι να κερδίζουν και οι δύο πλευρές. Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν να κάνουν εμπόριο με την Αφρική. Και βεβαίως ε, στην ασφάλεια έχουμε κάνει πολλά. Και χαιρόμαστε που τονίζετε την ε, διακυβέρνηση ότι πρέπει να αποκτήσει μια νομιμοποίηση η Αφρική μέσω μόνιμης θέσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας με τις ιδιαιτερότητές της. Ψάχνουμε ως Αφρικανική Ένωση για να δούμε πώς με συνέπεια μπορούμε να ε, συνεργαστούμε με όλους μας τους εταίρους. Και οι στόχοι που επιδιώκουμε είναι αυτοί που είναι στο θεματολόγιο μας για το 2063. Θεωρούμε ότι η Κίνα για μας είναι ένας από τους κύριους εταίρους. Στα πλαίσια, για παράδειγμα, της πολύμορφης ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη. Μας εντυπωσιάζει η ακρίβεια με την οποία απαντήσατε σε ερωτήσεις μας και η φιλοδοξία σας. για τις προοπτικές των σχέσεων της Αφρικανικής Ένωσης και της, ε, του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου με μας στα πλαίσια της ε, μετακοτονού εποχής. Ευχαριστώ πολύ. Και θα προεδρεύσει τώρα ο κύριος Ντέβα για το επόμενο σημείο. Παρακαλώ κύριε Ντέβα. Ευχαριστώ κύριε Λοπιθαγκυλάρ, λέει ο κύριος Ντέβα. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η συνέχιση που δόθηκε στο ψήσμα για το Εθνικό Πάρκο Βιρούγκα. Ιδιαίτερη κατάσταση ασφαλείας μετά την, ε, τα τραγικά, τα ιδιαίτερα τραγικά συμβάντα Θα πρέπει να συνδεθούμε τώρα με τον Εμμανουέλ Ντομεγόντ μέσω δορυφόρου και παρακαλώ τον κύριο Φρανσουά Ξαβιέ Ντονεά, υφυπουργό του Βελγίου, να έρθει στο Πρόεδρο.